Καλησπέρα σα. Ω συνήθω θα πρέπει να σα ενημερώσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται και μαγνητοσκοπείται. Μεταδίδεται μέσω διαδικτύου. Η ημερήσια διάταξη σας διανεμήθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2011. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, επιβεβαιώνεται ω έχει εκτός από το γεγονός ότι η Αντιπρόεδρος, η κυρία Γκουρμάη, δεν θα είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, επομένως δεν θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τη γνωμοδότησή της στο σημείο υπαριθμών 5 της ημερήσιας διάταξης και επομένως θα πρέπει να το αναβάλουμε για αύριο. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ενστάσεις, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση να σας κάνω, επομένως μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 που αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άσκηση του δικαιώματος έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντικατάσταση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19 Απριλίου του 1995. Η συγητής είναι ο κύριος David Μάρτιν. Του ζητώ να μας παρουσιάσει πώς έχει κατάσταση, να μας πει κατά πόσον κατατέθησαν και ποιε και αν υπάρχουν συμβιβαστικές τροπολογίε και να μας δώσει και κάποιες υποδείξεις για την ψηφοφορία. Παρακαλώ λοιπόν ο κύριος Μάρτιν να λάβει το λόγο. Um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχίζω ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους και για τις τροπολογίες, περίπου 30 που κατέθεσαν. Επίσης ευχαριστώ τη γραμματεία που όπως πάντοτε ήταν υπέροχη. Γιατί η έκθεση αυτή έχει αρκετή σημασία για το Κοινοβούλιο. Θα θυμάστε ίσως ότι δόθηκε νέα σημασία στο θέμα αυτό λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας. Τώρα έχει δικαίωμα πρωτοβουλία στο Κοινοβούλιο ως προς τους κανονισμούς για τη θέσπιση για προσωρινών επιτροπών έρευνας. Εδώ θα μιλήσω τώρα για τα όρια αυτής της δυνατότητας και θα προτείνω αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες ελπίζοντας να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες να φτάνουμε έτσι στην αλήθεια με τέτοιου είδους έρευνες. Η τελευταία τέτοια επιτροπή έρευνας έκανε και αυτή ορισμένες συστάσεις ως προς το πώς θα μπορούσε να ενδυναμωθεί η δικαιοδοσία του Κοινοβουλίου στο δικαίωμα έρευνας. Συμφωνείτε φαντάζομαι ότι και αυτή η έκθεση συμπεριλαμβάνει πλήρως εκείνες τις συστάσεις. Επίσης είχα λάβει υπόψη μου δύο άλλα σημαντικά σημαντικές προϋποθέσεις. Πρώτον, μία μελέτη που συνέκρινε την κατάσταση στις χώρες μέλη ως προς τα δικαιώματα έρευνας που έχουν οι χώρες για να είναι βέβαιο ότι δεν θα επικαλύπτει τις εθνικές δικαιοδοσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεύτερον, είχαμε λάβει πριν γράψω την έκθεσή μου And I also point that we've now got some draft compromises. προηγούμενες προτάσεις συμβιβασμού που είχαν γίνει με τη βοήθεια της νομικής υπηρεσίας. Σας υπενθυμίζω λοιπόν τις αλλαγές που προτείνω. Περισσότερες δικαιοδοσίε στις επιτροπές έρευνας για να διατάσσουν έρευνε, με πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έρευνα που διαθέτουν οι χώρες μέλη, τα ενωσιακά όργανα και φυσικά οι νομικά πρόσωπα. Πρέπει να έχει το δικαίωμα να καλεί, να εγκαλεί οι αξιωματούχους ή πολίτες ώστε για να απαντήσουν σε ερωτήσεις να ζητήσει μαρτυρίες και να ζητήσει από θεσμικά όργανα να δουν εκείνα, να εξετάσουν εκείνα ορισμένα άτομα. Το αίτημα κατάθεσης πρέπει να γίνεται σεβαστό από όποιον ζητηθεί και θα υπάρξουν κυρώσεις εφόσον διαπιστώνονται παραβιάσεις και τότε τα κράτη-μέλη θα λαμβάνουν δράση σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία. Για τα μέλη φοβάμαι ότι πρέπει αντί να τα πω ένα-ένα να τα πω γενικότερα. Ακόμη μια φορά ευχαριστώ τους συναδέλφους που κατέχασαν γιατί μερικές με βοηθάνε να αποσαφηνίσω ορισμένες πτυχές ιδιαίτερα ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον τονισμό του διαχωρισμού των εξουσιών με, του κάθε οργάνου. Μερικοί συνάδελφοι προσπάθησαν να το ενδυναμώσουν αυτό που εγώ όμως νόμιζα ότι ήδη το είχα συμπεριλάβει, αλλά τέλος πάντων το δέχομαι γιατί ξεκαθαρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστήριο και ότι ο ρόλος μιας προσωρινής Επιτροπής Έρευνας είναι να ξεσκεπάσει την αλήθεια. Τα αποτελέσματα δεν προβλέπονται, τα οι που θα επιβληθούν δηλαδή. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα πει ρητά, αλλά τέλος πάντων ας τα πούμε πιο σαφώς. Επίσης, στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών είναι ο βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης αυτής για να πετύχει αυτή στο μέλλον. Και αυτές οι τροπολογίες με βρίσκουν σύμφωνο. Ο κανονισμός του Κοινοβουλίου βέβαια πρέπει να προσαρμοστεί για να προβλεφθούν όλα αυτά και ευχαριστώ τους συναδέλφους που ζήτησαν και εκείνη η αλλαγή του κανονισμού. Αλλά δεν θέλουμε το διαθεσμικό αυτοκείμενο να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες για την εργασία του Κοινοβουλίου συγκεκριμένα μόνο. Θα χρειαστούν χωριστές εκθέσεις γι' αυτό μερικές από τις προτάσεις του κυρίου Βάιλα του ζητώ να μην συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ την έκθεση αλλά σε κάποια άλλη προσθήκη στον κανονισμό ή από σε οτιδήποτε προκύψει από τη διαθεσμική σχετική συμφωνία. Γενικά δέχομαι αν και δεν είναι όλοι οι συντάξει των προϊόντων εδώ, όλες τις τροπολογίες του κ. Βίλαν είτε πρόκειται για συμβιβασμού είτε όχι, όταν δεν αφορούν όμως τον εσωτερικό κανονισμό. Γενικά τις δέχομαι, μία-δύο θα ήθελα να τις ξανασυζητήσω με εκείνον, αλλά απορρίπτομαι όλες τις τροπολογίες του κυρίου Φόξ, εκτός από τις γλωσσικές, γιατί μας αφήνουν, αν γίνουν δεκτές, με το status quo, χωρίς καμία αλλαγή. Ενώ ο στόχος μας ακριβώς ήταν να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Φυσικά, Πρόεδρε, επειδή μόλις προσήλθαν πριν από μισή ώρα, δεν πρόλαβα να κάνω τους απαραίτητους συνδυασμούς και κατάλογο λεπτομερή των προτάσεων μου για τις τροπολογίες, αλλά θα το πράξω. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις για αυτά που σας είπα, νομίζω ότι θα προλάβουμε να συνάψουμε συμφωνίες και να ψηφίσουμε μέχρι αύριο. Θέλει να παρέμβει. Ο Παρακαλώ κύριε Είχε ζητήσει πρώτα το λόγο ο κύριος Νταφ, επομένως ε, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Νταφ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μάρτιν ε, για τα όσα έκανε για το θέμα αυτό, διότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι ακόμα δεν μας έχει δώσει ένα κατάλογο ψηφοφοριών. Δεν ε, νιώθει λοιπόν κανείς από εμά προετοιμασμένος να ψηφίσει αύριο το πρωί. Δεν είμαι αντίθετο στο να ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω δύο-τρία πράγματα σήμερα το απόγευμα αν γίνεται. Καταρχάς, Ο Επίτροπος Σεύκοβιτς απάντησε με σχόλια στο σχέδιο κειμένου και ο εισηγητής έλαβε υπόψη αρκετά από τα σχόλιά του. Θα μπορούσαμε ίσως να ακολουθήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι σε όλα τα θέματα, σε καμία περίπτωση, διότι θεωρώ ότι, ότι είναι πολύ αρνητική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Αλλά στο άρθρο 6.2, όπου η Επιτροπή επισημαίνει τον κίνδυνο να συμπεριλάβουμε και τα εμπορικά συμφέροντα για τα μελλοντικά στοιχεία στην ε, ε, δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν ένα μάρτυρα, θα πρέπει να είμαστε ίσως λίγο πιο προσεκτικοί και να συμπεριλάβουμε και την ε, προηγούμενη ρήτρα που έχουμε για τα εμπορικά συμφέροντα στο τέλος αυτής της φράσης. Διότι γνωρίζουμε ότι θα είναι αδύνατον ή τουλάχιστον απίθανο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διευκρινίσει ή να καθορίσει επακριβώς ποια είναι τα εμπορικά συμφέροντα σε κάποιες περιπτώσεις. Δεύτερον, για την παράγραφο 10 στην παράγραφο 10 λέμε ότι η Εξεταστική Επιτροπή θα μπορεί να διεξάγει επιτόπιες έρευνες. αλλά τα μέσα για τη διενέργεια των ερευνών αυτών είναι αποκλειστικά στα χέρια των εθνικών αρχών και υποψιάζομαι ότι είναι αποκλειστικά στα χέρια των εθνικών κοινοβουλίων. Και δεν είμαι βέβαιος κατά πόσον έχουμε ακόμα καθορίσει τις συστηματικές μας σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια επί του θέματος. Κάτι τέτοιο θα διευκολύνει ίσως τις έρευνές μας. Ίσως θα πρέπει να γίνει μια επίσημη ε, συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια επί του θέματος αυτού, ώστε να διαπιστώσουμε μέχρι ποιου σημείο είναι και διατεθειμένοι αλλά και ικανοί να φτάσουν. Mm-hmm. όσον αφορά μια εξεταστική επιτροπή ε, έρευνας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρθρο 17. Ένας σημείο σημασίας. Ε, το σημείο 17.3 θα το διέγραφα, διότι νομίζω ότι ουσιαστικά προτρέπει έναν εμπειρογνώμονα να μας υποδείξει κάποιο δυνητικό μάρτυρα και δεν ξέρω αν είναι σωστό να υπάρχει τέτοιο δέλεαρ για τους εμπειρογνώμονες. Τέλος, Και εδώ είναι θέμα πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Το πρώτο τμήμα στο άρθρο 1 προσπαθούμε να καθορίσουμε ποιο είναι το αντικείμενό μας. Στην πράξη, Ένα από τα πολύ σημαντικά σημεία της συνθήκης λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δράσει μόνο βάσει των καθηκόντων του και των αρμοδιοτήτων του. Και επειδή αυτό υπάρχει στο άρθρο 2, στη σύσταση και εντολή εξεταστικών επιτροπών, νομίζω ότι θα πρέπει να αν το εξετάσουμε λίγο καλύτερα, καλό θα ήταν να αναφέρεται στο άρθρο 1. Διότι το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού αφορά τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι της αρεσκίας μας. Και νομίζω ότι ε, θα προσδώσει περαιτέρω νομική σαφήνεια το οποίο θα είναι και αυτό το οποίο κανονικά πρέπει να κάνουμε. προκειμένου να αντικατοπτρίζεται και πλήρως η συνθήκη στο πρώτο άρθρο του κανονισμού αυτού. Αν μεταφέρουμε λοιπόν το σημείο αυτό από το άρθρο 2 στο άρθρο 1. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ κύριε Νταφ. Ο κύριος Χέφνερ έχει το λόγο. Σε Ευχαριστώ Πρόεδρε και από πλευρά μου συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Μάρτιν. Σας ευχαριστώ για την πολύ καλή πρόταση. Προτού περάσω στις λεπτομέρειες και στις μεμονωμένες τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, να πω κάτι επί της αρχής. Να κάνω μια γενική παρατήρηση και σε ό,τι αφορά την επιστολή του Επιτρόπου Σεύκοβιτς, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα και τον οποίο θεωρώ ιδιαίτερα σοβαρό, ωστόσο θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να τον ακολουθήσουμε σε όλα όσα προτείνει. Θεωρώ επίσης ότι η θέση της νομικής μας υπηρεσίας σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού μας για τα δικαιώματα των εξαστικών επιτροπών του Κοινοβουλίου είναι πιο σωστές οι προτάσεις αυτές και ότι το άρθρο 326 ε, της ε, Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εφαρμογή. Τα θέματα αυτά δεν μπορεί να επιλύονται στα κρατη Μιλάμε για πολλές αδυναμίες για την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου και εδώ έχει αρμοδιότητα με καλύτερη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτά που θεωρώ ότι αποτυπώνονται στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θεωρώ και υποστηρίζω τη θέση του εισηγητή και της έκθεσης και θεωρώ επίσης ότι τα θέματα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όπου υπάρχουν διστάμενες απόψεις, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τα οποία συντείνουν στο να υποστηριχθεί η θέση της έκθεσης και του εισηγητή. Τώρα, εν συντομία να περάσω σε κάποια μεμονωμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες. Τη κυρία Γιαννάκου τη Τροπολογία, τη υποστηρίζω και τις δύο. Θεωρώ ότι είναι σαφέ και αυτονόητο δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε γιατί. Δυσκολεύομαι και ίσως να με βοηθήσει η παρουσίαση της κυρίας Γιατεμέκη. Δυσκολεύομαι με τις τροπολογίες της Μίλα για τις κυρώσεις και το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι δικαστήριο. Μα δεν είπε κάτι τέτοιο ο οι κυρώσει δεν επιβάλλονται μόνο από δικαστηρία και αστυνομία, για παράδειγμα, μπορεί να επιβάλλει κάποιε κυρώσει. Και σε κάποιε χώρε υπάρχει η δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσει από εξεταστικέ επιτροπέ. Και θεωρώ ότι όλα αυτά δικαιολογούνται από το άρθρο 229 της συνθήκης Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσετε με καλύτερο τρόπο τι εννοείτε. Ε, Ιδάλλως δεν μπορώ να συμφωνήσω με την τροπολογία στην παρούσα μορφή της για τις προτάσεις του, προτάσεις του κυρίου Βίλαντ τώρα. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση συμφωνώ με όλες αυτές τις ε, τροπολογίες. Πολύ σημαντικό φαίνεται να είναι το θέμα της ε, ψήφου μειοψηφία ε, μια εξεταστική επιτροπή. Γιατί η εμπειρία καταδεικνύει ότι υπάρχουν καταστάσει κατά τι οποίε δεν συμφωνούν όλα τα μέρη του Κοινοβουλίου, του κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τις εξεταστικές επιτροπές, γιατί μπορεί η διαπίστωση των ε, γεγονότων να γίνει καταρχάς με ψήφο μειοψηφίας. Νομίζω ότι και αυτό θα έπρεπε να καταστεί πρακτική. Και να ρωτήσω τον κύριο Βίλαντ το 1 τέταρτο των προτάσεων του. Αν θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν συγκρίσιμες και προβλέπονται συγκρίσιμες περιπτώσεις ε, από τον κανονισμό σε ό,τι αφορά την ε, συγκέντρωση του ενός τετάρτου όλες οι τροπολογίες του κυρίου Φόξ ε, έχουν να κάνουν με την αποδυνάμωση των εργαλείων μιας τέτοιας εξαστικής επιτροπής. Μα δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι θα συνέφερε τον κύριο Φόξ αν υπάρχει κάποια παρανόηση, κάποια σύγχυση, να υπάρχουν δυνατά εργαλεία για να ερευνηθεί. Άρα δεν συμφωνώ με την πρόταση αυτή του κυρίου Φόξ. Και κλείνοντας, να ρωτήσω τον κύριο Βίλα για την τροπολογία 27. Γιατί συμφωνώ, σας είπαμε σχεδόν όλες τις τροπολογίες σας, αλλά εδώ πέρα δεν έχω αποφασίσει, γιατί θεωρώ ότι υποδυναμώνεται το κείμενο. Σε σχέση με αυτά που προτείνει ο εισήγητη. Ιδιαίτερα γιατί υπάρχουν και κάποιες χώρε όπου δεν υπάρχει καν ε, πρόβλεψη κυρώσεων. Δηλαδή, αν λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προσανατολισμό στο σύστημα κυρώσεων που προβλέπεται από τα κράτη-μέλη, είναι πάρα πολύ, διάστατα τα πράγματα ανάλογα με το κράτο μέλο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο σαφείς. Καταλαβαίνω φυσικά ποια είναι το νομικό υπόβαθρο από κάτω που μας προκαλεί προβλήματα, αλλά Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω με την καλή, για την καλή έκθεση, για την καλή δουλειά που κάνατε. Ακόμα και αν περάσουν κάποιες τροπολογίες, θεωρώ ότι επί της αρχής έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και ότι πρέπει να προβάλλουμε αυτή την άποψη στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ε, ο κύριος Βίλαντ έχει ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και συγγνώμη που καθυστέρησα. Χάρηκα που άκουσα τα ευγενικά σχόλια του κυρίου Χέφνερ και μου είπαν και την, τι είπε ο κύριος ε, Μάρτιν. Έχω δύο βασικά στοιχεία τα οποία ήθελα να αναφέρω. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Και να απαντήσω και στον κύριο Χέφνερ. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη μειοψηφική ψήφο, θεωρώ ότι υπάρχει ένα μασικό στοιχείο. Μιλάμε για την τροπολογία υπαριθμών 13, όχι συγγνώμη λέει ο Η 13. Στην οποία δεν συμπεριέλαβε η συμβαστική πρόταση του κυρίου Μάρτιν. Αυτό θεωρώ ότι είναι βασικό. Έχει να κάνει με τις ε, μειοψηφικές ψήφους. Δεν μπορώ να φανταστώ να κάνουμε μία εκτενή εργασία Εξεταστικής Επιτροπής. Και τελικά, τι θα γίνει με αυτά τα κείμενα. Θα ήθελα λοιπόν να βρω ένα τέτοιο, μια τέτοια λύση. Είτε η Ολομέλεια θα απορρίψει και τα δύο τμήματα και δεν θα υπάρξει συμπέρασμα της ε, Εξεταστικής Επιτροπής ή θα σημειωθούν και οι δύο απόψεις. Εγώ λοιπόν θα επιμείνω σε όλα αυτά που αναφέρονται στην τροπολογία επαριθμό 13. Νομίζω ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα αποδυναμωθεί αν μετά από μια ε, εξαστική επιτροπή διαφωνήσουμε για παράδειγμα για κάποιο κόμμα ή κάποια τελεία και τελικά αποδυναμωθεί η έκθεση της Εξεταστικής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία αυτή, την μειοψηφική αυτή ψήφο. Νομίζω ότι όσοι δεν είναι παρόντες δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα εφόσον δεν έχουν αγωνιστεί και αυτοί. Άρα θεωρώ ότι η απαρτία του ενός τετάρτου είναι λογική ουσία λοιπόν αυτής της απαρτίας είναι κάτι το οποίο χρήσει αντικειμενικότητας. Αυτή λοιπόν η διπλή πρόβλεψη του 5% σε ό,τι αφορά και την ολομέλεια. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 27 που μου θέσατε την ερώτηση εξηγήθηκε ότι είναι δικαίωμα της Εξαστικής Επιτροπής και εμείς έχουμε τη δυνατότητα από το πρωτογενές δίκαιο να προβλέψουμε και κάποιες κυρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν αναφέρω ότι το ελάχιστο το οποίο θέλω να πετύχω να υπάρχουν ανάλογες κυρώσεις τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται στο εκάστοτε κρατός μέλος. Γι' αυτό λοιπόν θέλω τα κράτη-μέλη να δεσμευθούν σε περίπτωση παροβιάσεων, σε περίπτωση ε, σφαλμάτων στο ποινικό τους δίκαιο, να προβλέπουν αρμοδιότητες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση που πρέπει να εισαχθεί με το κείμενο αυτό και περνάω στο τελευταίο σημείο τώρα. Επιμένω ότι δεν είναι στην ελεύθερη διακριτική ευχαίρεια ενό ε, μάρτυρα κατά πόσον δημόσια ή μη δημόσια ορκωτά ή μη ορκωτά θα καταθέσει. Αυτό εξαρτάται από την Εξαρτική Επιστροπή. Και αν αυτό κάπως λίγο τρομάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν μπορούμε προς τα έξω να ζητάμε διαφάνεια. Και να διοργανώνουμε άψογα τέτοιες διαδικασίες και μετά να λέμε ότι θα εξαρτάται από την επιτροπή αυτή κατά πόσο θα γίνει δημόσια ή μη η κατάθεση ενός μάρτυρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν θεσμικές συνέπειες και δυσκολίες. Εγώ θα ήμουν διατεθειμένος μαζί με τον συνάδελφο Μάρτι να τα ψηφίσουμε όλα αυτά αύριο και να βγούμε στην Ολομέλεια και να εξηγήσουμε πριν από την ψηφοφορία να κάνουμε διαπραγματεύσεις και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να καταδείξουμε ότι στο θέμα του πώς καταθέτουν οι μάρτυρες να πούμε ότι για παράδειγμα για την ε, πρόταση αυτή του κυρίου Μάρτιν έχουν κατατεθεί 500-600 ψήφοι για να αποτελεί και αυτό ένα πολιτικό βάρος και να επανέλθουμε πάλι με την έκθεση αυτή και με την πρόταση αυτή στην Ολομέλεια. Mm. Allora, visto che non επειδή δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να έχουν ζητήσει το λόγο, θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Αναστασόπουλο, να μας ε, πει την άποψή του για τα όσα άκουσε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναστασόπουλος ήταν το όνομα ενός πολύ γνωστού κοινοβουλευτικού εγώ έχω μια συλλαβή λιγότερο Αναστόπουλος λέγομαι, Αναστόπουλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να εκφραστώ εδώ μέσα πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Ο Αντιπρόεδρος Εύτσεβιτς, όπως υπόθηκε ήδη, μπόρεσε ήδη να συμμεριστεί με τον εισηγητή αλλά και άλλα μέλη της Επιτροπής σας μέσω της Γραμματείας τις σκέψεις του ή και τις ανησυχίες του ακόμη αλλά όπως λέει και η επιστολή του αυτά όλα με επικοδομητικό πνεύμα γιατί η Κομισιόν θέλει με επικοδομητικό πνεύμα να συμβάλλει. Φυσικά εδώ βρισκόμαστε σε διαδικασία σύμφωνης γνώμης και γι' αυτό η Κομισιόν θα μπορέσει επίσημα να εκφραστεί αφού το Κοινοβούλιο υποβάλει την πρότασή του, κάνει τη γνωμοδότησή του. Θα δούμε τι θα πούμε, υπέρ ή κατά, αλλά δεν φτάσαμε ακόμη εκεί. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μιλήσω για τρία σημεία της εκθέση αυτής που ανέφερε ένα προς ένα ο Αντιπρόεδρος. Καλό θα ήταν νομίζω να αποσαφηνίσουμε στο πρώτο άρθρο, στο πρώτο σημείο, ότι εδώ ισχύει το 226, το οποίο μιλάει για ένα πλαίσιο άσκησης της εντολής του Κοινοβουλίου. Τι εννοεί αυτό ακριβώς. Γιατί στο ίδιο άρθρο επίσης λέει ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς να αποκλείεται διαβούλευση και με άλλα όργανα για να μην υπάρξουν προβλήματα λοιπόν νομίζουμε ότι πρέπει να ορίζεται έτσι σαφέστερα ποιο είναι το εύρο στο πεδίο εφαρμογής και αφού καθοριστεί καλύτερα αυτό στο πρώτο σημείο και τα υπόλοιπα μετά θα φωτιστούν από αυτό το φως, το 10, το 11, το σημείο για το πώς θα γίνονται οι καταθέσεις, πώς θα υποβάλλονται οι αιτήσει για υποβολή εγγράφων, Όλα αυτά θα απορρέουν από, αυτήν, από αυτόν τον καλύτερο, σαφέστερο ορισμό του πεδίου εφαρμογής. Δεύτερον, το σημείο 15 που αφορά τις μαρτυρίες των υπαλλήλων, τους υπαλλήλους που καλούνται να καταθέσουν. Εδώ πρέπει να προσέξουμε γιατί αυτά που προβλέπει ένας κανονισμός σύμφωνα με το 226 δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση με κανονισμούς που θα βασίζονται στο 336 της συνθήκης που αφορά το, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων και όπου ορίζεται ρητά ποια είναι τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Υπάρχει και ένα πρόσφατο έγγραφο για το καταστατικό του διαμεσολαβητού που αποτέλεσε και αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων και όπου ορίζεται ακριβώς πώς μπορεί να δώσει μαρτυρία ένας υπάλληλος. Τέλος, τρίτον, οι κυρώσεις, το σημείο 18 πρέπει να προσέξουμε το εξή εδώ. Ένας κανονισμός παραγόγου δικαίου δεν πρέπει να αντιφάσκει με το πρωτογενές δικαίου. Και εννοώ το πρωτόκολλο που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υπαλλήλων. Αυτά όλα τα λέμε για να βοηθήσουμε, να σας βοηθήσουμε στην ανάλυση σας. Θα είμαστε παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της ανάλυσης σας. Προς στιγμή δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα γιατί δεν έχουμε ακόμη μπροστά μας το επίσημο κείμενο του Κενοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αναστόπουλο. Το είπα σωστά το όνομά σας τώρα. Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλες παραμβάσεις, οπότε να ζητήσω από τον συνάδελφο τον κύριο Μάρτιν να σχολιάσει τα όσα ακούσαμε και επίσης να αποφασίσουμε αν είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε αύριο το πρωί που νόμιζα ότι ήταν αυτό που είχε ζητήσει και ο κύριος Μάρτιν ή εάν θα μπορούσαμε να αναβάλουμε και για κάποια άλλη ημερομηνία όπως και να έχει πριν από τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου, δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου. Θα αποφασίσουμε ε, και θα μας πει την άποψή του και ο εισηγητής, ε, αφού σχολιάσει τα όσα άκουσε. Καταρχάς, για το θέμα της ψηφοφορίας. Κύριε Πρόεδρε, η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην ψηφίσουμε αύριο. Ο κύριος Βίλαντ έπρεπε να φύγει, αλλά νομίζω ότι με τα χαρά θα μπορούσε να ψηφίσει. Ε, η ομάδα μου δεν έχει πρόβλημα. Δεν θα υπάρχει απόλυτη συνένεση βέβαια, αλλά νομίζω ότι μέχρι εδώ μπορεί να φτάσει η συνένεση την οποία θα καταλήξουμε. Με περαιτέρω συζήτηση δεν νομίζω ότι θα επιτύχουμε και πολλά περισσότερα. Και θα ήθελα να πω και σε όλους τους συναδέλφους ότι ό,τι και να εγκρίνουμε είτε εδώ είτε στην Ολομέλεια ε, εξαρτάται και από το τι θα κάνει από εκεί και πέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί είναι μόνο το πρώτο στάδιο. Μετά θα πρέπει να κάνουμε διοργανικές συζητήσεις. Αυτό που προτείνω είναι να βγει όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα εδώ από την Επιτροπή μας και να ακούσουμε από εκεί και πέρα τι έχουμε να κάνουμε με άλλα όργανα. Αλλά ούτως ή άλλως, αν ξεκινήσουμε συζήτηση με άλλα όργανα του Ευρωπα... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε. Είμαστε στην αρχή της διαδικασίας λοιπόν, αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε φιλόδοξα. Επίσης να πω, επειδή το ανέφεραν και οι τρεις ομιλητές, ότι ε, χαίρομαι για τη συνεργασία με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Ε, δική μου πρωτοβουλία ήταν η πρώτη συνάντηση. Η επιστολή του, παρά το γεγονός ότι δεν με βρήκε σύμφωνο σε όλα τα σημεία, ήταν πολύ επικοδομητική και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καρποφόρο διάλογο, κάτι το οποίο με χαροποιεί ιδιαίτερα. Τώρα, ε, για τα σχόλια του κυρίου Νταφ. Το σχόλιο του για το άρθρο 6.2 νομίζω ότι πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα αποτανθώ και στην νομική υπηρεσία για να δω ε, κατά πόσον μπορούμε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν νομίζω όμως ότι είναι κάτι που δεν μπορούμε να λύσουμε και σε κατοπινό στάδιο, αν ε, δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Για το άρθρο 10 όμως, διαφωνώ με τα σχόλιά σας εύλογο το επιχείρημα ότι δεν είμαστε εθνικό κοινοβούλιο και επομένω δεν μπορούμε να επιβάλλουμε τα ίδια πράγματα για τι εξεταστικές επιτροπέ που τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά αν δείτε την ε, σχετική τροπολογία που έχουμε εδώ, την οποία θα υποστηρίξω, ε, για να έχουμε ε, κοινή εξεταστική έρευνα με τα εθνικά κοινοβούλια, θα διευκρινιστεί πολύ περισσότερο το θέμα αυτό. Αν διαβάσετε δε και το άρθρο αυτό, ε, στο πλαίσιο και των υπολείπων άρθρων, είναι σαφές ότι το δικαίωμα να διαρεγνούνται επιτόπιες έρευνας είναι περιορισμένο και μόνο όταν θεωρεί η Εξεταστική Επιτροπή ότι μπορεί να εκλάβει στοιχεία τα οποία απαιτούνται για να διαμορφώσει άποψη και να λάβει απόφαση. Αν το εξετάσουμε μεμονωμένα, βεβαίως φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει έρευνες ε, χωρίς ε, να υπάρχει λόγος και να είναι στο το κράτος μέλος κλπ. Δεν είναι αυτό το νόημα και δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε εδώ. Ε, στο άρθρο 17.3 τώρα, αυτό το βασίσαμε σε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και απλώς ε, μεταφέρουμε την απόφαση εδώ στο κανονισμό. Νομίζω ότι υπερερμηνεύουμε αυτό που σημαίνει στην πράξη. Δεν σημαίνει ότι θα καλούμε έναν πυρογνώμονα και θα του ε, λέμε να ε, μας υποδείξει μάρτυρες ή να επιλέξει μάρτυρες. Μας λέει απλώς ποιοι είναι πιθανόν. Δεν μας λέει να μιλήσετε με τον Τάδε γιατί κάτι κρύβει. Απλώς μας υποδεικνύει τι ακριβώς θα μπορούσαμε να κάνουμε στην έρευνα. Δεν ξέρω αν το εξήγησα πολύ καλά, αλλά είναι κάτι διαφορετικό και εγώ το βλέπω κάπως έτσι. Η παρατηρήση τώρα του κυρίου Χέφνερ. Αναφερθήκατε στι ε, τροπολογίες της κυρίας Γιαννάκου Υπάρχουν κάποιες συμβαστικές προτάσεις οι οποίες θα παρουσιαστούν είτε αργότερα σήμερα είτε αύριο και νομίζω ότι θα σας ικανοποιήσουν οι συμβαστικές τροπολογίες. Για την τροπολογία της κυρίας Γιατρυμάκη συμφωνώ με την ανησυχία σας για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχουμε συμφωνήσει σε μια συμβαστική πρόταση η οποία δεν με ικανοποιεί κατά 100% ότι δέχτηκα εν είδη συμβιβασμό, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό να το βρω. Δεν το βρίσκω. Δεν το βρίσκω. λέει ότι το δόγμα του διαχωρισμού ε, αρμοδιοτήτων θα πρέπει να γίνει σεβαστό όταν ε, ε, γίνεται κατάφρηση από το νομοθετικό, δηλαδή το κοινοβούλιο, το εκτελεστικό, δηλαδή κυβέρνηση και το δικαστικό, δηλαδή το δικαστήριο, θα είναι ξεχωριστά και διαγράφεται η τελευταία φράση. Για μένα είναι περιττό, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά εάν καθησυχάσει τους πάντες, ε, το να το συμπεριλάβουμε δεν κάνει και κανένα κακό, αν μου επιτρέπετε να το θέσω έτσι. Δεν κάνει και πολύ καλό, αλλά σίγουρα δεν βλάπτει κανένα. Τροπολογία 27 όπου διαφωνούν οι κύριοι Χέφνερ και Βίλαντ, εγώ είμαι διατεθειμένο να δεχτώ την τροπολογία του κυρίου Βίλαντ, διότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα που έχουμε. Ο μόνο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικέ κυρώσει είναι μέσω ε, των παροστών διαδικασιών, δηλαδή των Εθνικών Κοινοβουλίων, και υπ' αυτό το πνεύμα δέχτηκα την ε, ε, τροπολογία. Τώρα, για τι παρατηρήσει του κυρίου Βίλαντ. Συμφωνώ με την τροπολογία 13 του κυρίου Βίλαντ, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να τίθεται τέτοιο θέμα σε διπηρεσιακή συμφωνία. Όταν θα καταλήξουμε σε διπηρεσιακή συμφωνία, όπω σα είπα και προηγουμένω, θα πρέπει να αλλάξουν ο κανονισμό του Κοινοβουλίου. Επομένω να δεχτούμε κάτι ε, το οποίο μπορεί και να αλλάξει τον κανονισμό του δικαστηρίου, αλλά δεν θα πρέπει να το κάνουμε μόνο και μόνο για να καταλήξουμε σε συμφωνία, διότι για να καταλήξουμε σε διοργανική συμφωνία θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα όργανα. Η τροπολογία 13 λοιπόν και μία ακόμα εργα... Ε, τροπολογία της οποίας ο αριθμός μου διαφεύγει που αναφέρει το ποσοστό που απαιτείται για μειοψηφική άποψη νομίζω ότι απαιτούν αλλαγή του κανονισμού του Κοινοβουλίου και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει πρώτα με τη διοργανική συμφωνία. Για την ε, τροπολογία 27 που ανέφερε ο κύριος Βίλαντ, εγώ το σκέφτηκα και με τους συμβούλες μου και δεν μπορούσαμε να αποφασίσουμε επ' αυτής, αλλά αφορά η τροπολογία 27 το κατά πόσο μπορεί να γίνει και κλεισμένο των θηρών μία συνεδρίαση εάν το ζητήσουν οι μάρτυρες. Έχει δίκιο ο κύριο Βίλαντ. Ναι. Μπορεί να υπάρχουν κάποιε περιπτώσει όπου θα πρέπει να γίνει συνεδρία και των θυρών και θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα επιλογή να πούμε όχι, θα γίνει δημοσίω. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε σάλ εδώ και όχι μέη και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστότερη διατύπωση και μπορώ να τη δεχτώ και αυτήν ε, την τροπολογία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Α, ναι. συγγνώμη, το άρθρο 1, το άρθρο 1. Κατανοώ τι λες, Άνδριο, ακριβώς Αν μου δώσει μια προφορική τροπολογία απόψε, θα προσπαθήσω να τη συμπεριλάβω αύριο στα όσα θα ψηφίσουμε. Ο κύριο Ντάφ θέλει το λόγο μετά από τη διευκρίνηση. Όχι, ωραία. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε με το σημείο αυτό τη συζήτηση και να πούμε ότι αύριο το πρωί θα γίνει η ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Μάρτιν για την ε, πολύ εύστοχη εκθεσή του και για τα όσα έκανε και περνάμε στο σημείο υπαριθμών 4, αναθεώρηση του άρθρου 70 του κανονισμού, που αφορά τις διαπραγματεύσεις στα πλαίσια μιας νομοθετικής διαδικασίας σε διοργανικό επίπεδο. Το γραφείο της Προεδρίας ε, κάλεσε την Επιτροπή μας να επανεξετάσει το άρθρο 70, το οποίο έχει σχέση και με τον κώδικα διοντολογίας που θα συζητήσουμε ε, και υπάρχει μια επιστολή που μας ζητά γνωμοδότηση και μας ζητά αν πρέπει να είναι περισσότερο δεσμευτικές οι υποδείξεις που περιλαμβάνονται σήμερα στο σύστημα του άρθρου 70 και του κώδικα δεοντολογίας όπως προβλέπεται ε, στο παράρτημα υπαριθμών 20. Ο εισηγητή είναι ο κύριος Γκερέρο, ο οποίος έκανε έρευνα, μελέτε, ήρθε σε επαφή με κόσμο και θα μα παρουσιάσει σήμερα νομίζω ένα έγγραφο εργασία. Έχω δίκιο? Παρακαλώ κύριε Γκερέρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας πω λίγα πράγματα για το χρονοδιάγραμμα. Πώς σκοπεύω να ασχοληθώ με αυτό το ε, θέμα στο άρθρο 70, αναθεώρηση στο άρθρο 70. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο συνοδεύεται και με κάποιες συστάσεις οι οποίες έγιναν από τη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Στα τέλη Οκτωβρίου θα αποστείλω προς μετάφραση μία προσωρινή έκθεση, ένα σχέδιο έκθεσης, με στόχο να μπορέσουμε να συζητήσουμε αυτή αυτό το σχέδιο έκθεσης στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω διαμακρών τους λόγους για τους οποίους ζητήθηκε από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων να αναθεωρήσουμε το άρθρο 70 του κανονισμού και τι προβλήματα δημιουργούνται σε αυτή την αναθεώρηση και τις γενικότερες λύσεις που προσφέρονται σε αυτό το έγγραφο εργασίας προκειμένου να κάνουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η ουσία ξεκινάει από μία συζήτηση που έχουμε επανειλημμένως όταν υπάρχει μεγάλη νομοθετική δραστηριότητα σε ένα κοινοβούλιο όπως ακριβώς γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το θέμα λοιπόν είναι πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την εκπροσώπηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό και στην Ολομέλεια και ε, για τους ευρωβουλευτές άνδρες και γυναίκες αυτού του Κοινοβουλίου με την αποτελεσματικότητα στην νομοθετική διαδικασία και με την ικανότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις όταν δεν είναι ε, πολύ σοβαρά τα ζητήματα με απλουστευμένο τρόπο. Όπως ξέρουμε αυτές τις συζητήσεις τις κάνουμε και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Κάθε φορά που προσπαθούμε να διατηρούμε τη συνεδρίαση ομολομελία για τι πολιτικέ συζητήσει και τη συνεδρίαση τη Επιτροπές για την επίλυση των πιο τεχνικών, ε, διαδικαστικών ε, ή απλούστερων θεμάτων ε, στις νομοθετικές επιτροπές. Υπάρχει όμως ένα θέμα διαφάνειας. Και το κοινοβούλιο αυτό πρέπει να προχωρήσει στα πλαίσια της δημοκρατίας και στην δημοσιοποίηση των θεμάτων αυτών στην κοινή γνώμη. Το, η κοινή γνώμη πρέπει να γνωρίζει τι συζητά το Κοινοβούλιο, σε τι συμφωνίες καταλήγει το Κοινοβούλιο και θα πρέπει επίσης να συνειδητοποιεί ο, τι ακριβώς έκαναν οι εκπρόσωποι του στα πλαίσια όλης αυτής της διαδικασίας. Στην προηγούμενη θητεία εγκρίναμε ένα κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος ε, αποτελεί σήμερα το παράτημα 20 του κανονισμού μας και ο οποίος επιλύει την πλειονότητα των προβλημάτων που θα μπορούσαν να αφορούν τα θέματα της διαφάνειας. Το πρόβλημα όμως έγκυται στο γεγονός ότι ο κώδικας αυτός δεν έχει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα σε τέτοιο βαθμό όπως τον έχει ο κανονισμός περιλαμβάνει πάντα μία πολιτική εντολή, μία ηθική υποχρέωση από πλευράς αυτού που διαπραγματεύεται σε πρώτη ανάγνωση, αλλά δεν έχει νομικό υποχρεωτικό χαρακτήρα, που σημαίνει δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για το σκοπό αυτό στον κανονισμό. Και αυτή η δυσλειτουργία σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο εισηγητής ο οποίος έχει αναλάβει τη διαπραγμάτευση σε πρώτη ανάγνωση. τίμησε ή δεν τίμησε αυτό τον κώδικα διοδολογίας, συμπεριφέρθηκε βάσει των αρχών της διαφάνειας και της ευθύνης, αλλά όχι πάντα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, τόσο η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών σε πρώτο στάδιο και η διάσκεψη των Προέδρων συζήτησαν στο δεύτερο εξάμεινο του 2010 επανειλημμένο στο ζήτημα και ε, υιοθέτησαν κάποιες συστάσεις τις οποίες ε, ε, έφτασαν εδώ στην Επιτροπή μας το 2011. έγινε μια εξέταση των γεγονότων της πραγματικότητας και της εμπειρίας που έχουμε από την αρχή της ε, ε, κοινοβουλευτικής αυτής θητείας και η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών κατέληξε σε μια σειρά από συστάσεις τις οποίες ε, διαβιβάζω εγώ στους ε, συναδέλφους. Καταρχάς θεωρεί ότι η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση δεν γίνονται εις βάρος των δυνατοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο μπορεί να χρησιμοποιήσει μηχανισμούς πρώτης, δεύτερης ανάγνωσης, συνδιαλλαγής, μπορεί να ε, περιορίσει όλες τις, ε, να περάσει σε όλα τα στάδια μιας διαδικασίας, αλλά εάν καταλήξει σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αυτό δεν είναι εις βάρος της δυνατότητας παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ιδίω επειδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάντα τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του για το αποτέλεσμα μια συμφωνία ε, η μια διαπραγμάτευση Η απόφαση λοιπόν να προσπαθήσουμε προσπαθήσουμε τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ε, θα πρέπει να λαμβάνεται αναπερίπτωση. Δεν χρειάζεται να καταληξουμε σε κάποιος γενικός κανόνας, απλώς θα πρέπει να λαμβάνεται αναπερίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις ε, διαφορετικές προϋποθέσεις που ισχύουν, το κατά πόσον υπάρχει ε, διάσταση απόψεων ε, ως προς μία έκθεση, αν είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα, εάν περιλαμβάνεται στις νομοθετικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το ενδιαφέρον της ε, δεδομένης εκπεριτροπής προεδρίας για να καταλήξουμε σε συμφωνία νωρίτερα. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις προϋποθέσεις και βάσει αυτών, αναπερίπτωση, αποφασίζεται αν θα γίνει διαπραγμάτευση για συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ή όχι. Η διοργανική συμφωνία ε, στην οποία κατέληξε το Συμβούλιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο το 2010, ε, λέει ότι ή δυνατόν, εάν είναι εφικτό, θα πρέπει να καταλήγουμε σε απόφαση σε πρώτη ανάγνωση. Να σας δώσω και κάποια στατιστικά στοιχεία. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, το 72% των θεμάτων ολοκληρώθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, το 11% ε, στο λεγόμενο Erling Second Reading, στις αρχές της δεύτερης ανάγνωσης, ένα 10% ε, σε δεύτερη ανάγνωση και ένα 5% σε συνδιαλλαγή. Δηλαδή, τρία στα τέσσερα θέματα κατέληξαν σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και αυτό θεωρείται λοιπόν ότι είναι ένας απόλυτα λογικός και διάφανος ε, μηχανισμός. Μετά από αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς σας είπα ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ένα δυσοπίλητο ή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους χρειάζεται να γίνει μεταρρύθμιση ε, και αναθεώρηση συγγνώμη, του άρθρου 70. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Καταρχά η συμμετρία βάσει επιτροπών. Υπάρχουν κάποιε επιτροπέ που εφαρμόζουν με μεγάλη αυστηρότητα και πολύ σοβαρή δέσμευση τους, ε, τον κώδικα διοντολογία και υπάρχουν και κάποιε άλλε επιτροπέ που δεν το κάνουν με την ίδια αποφασιστικότητα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πάντα σαφής η διαπραγματευτική εντολή για κάθε επιτροπή. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει μια εντολή με κάποιες γενικές ε, κατευθύνσεις, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψη μια εντολή σε μια έκθεση η οποία εγκρίθηκε με τις τροπολογίες οι οποίες πέρασαν στη συγκεκριμένη επιτροπή. Ναι. Δεύτερον, δεν διαβιβάζονται πάντα πληροφορίες στους σκιώδεις εισηγητές για το πώς ε, πάει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, της τριμερής συνομιλίας δεν προσκαλούνται πάντα ή δεν προσκαλούνται γέρος. Ε, δεν τους δίνεται πάντα η απαραίτητη τεκμηρίωση προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Και αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι δεν είναι πολύ συχνές, ο εισηγητής ε, έχει ένα επίπεδο αυτονομίας και ανεξαρτησίας που είναι εις βάρος του κοινού συμφέροντος της αρμόδιας επιτροπής και λίγο πολύ κάνει τα δικά του. Τέταρτο και πέμπτον, η αρμόδια επιτροπή συχνά δεν έχει περισσότερες πληροφορίες από την ε, διαπραγματευτική διαδικασία μέχρι το σημείο στο οποίο καταλήγουμε σε συμφωνία. Ε, ορισμένες φορές αφού καταλήξουμε σε συμφωνία τότε ενημερώνεται η αρμόδια επιτροπή. Και υπάρχει και κάτι το οποίο σίγουρα γνωρίζουν και οι βουλευτές και το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, γνωρίζουν πολύ καλύτερα από μένα. Ορισμένες φορές δεν υπάρχει αρκετός χρόνος από τη στιγμή στην οποία εγκρίνεται κάτι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τη στιγμή στην οποία γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια και δεν υπάρχει χρόνος για συζήτηση στις πολιτικές ομάδες και για να προετοιμάσουν την κοινή τους θέση στην Ολομέλεια. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τα προβλήματα αυτά, όπως είπε και ο πρόεδρος στην εισαγωγή του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέστειλε μια επιστολή στον κύριο Καζίνη ζητώντας η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων αφενός να εξετάσει την πιθανή αναθεώρηση του άρθρου 70 του κανονισμού, καθώς επίσης και καθορίζοντας και κάποια σημεία τα οποία ίσως θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για αυτή την αναθεώρηση. Μεταξύ αυτών τα εξής. κάποια σημεία τα οποία βρίσκονται στον κώδικα διοντολογία και τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά θα μπορούσαν ίσως να μεταφερθούν στο διατακτικό του άρθρου 70 και να γίνουν λοιπόν υποχρεωτικής φύσεως για τους ευρωβουλευτές. Υπάρχουν τέσσερα θέματα τα οποία αναφέρονται στην επιστολή αυτή που αποτελούν και την ουσία της υπόθεσης. Καταρχάς, Η απόφαση να γίνει διαπραγμάτευση σε πρώτη ανάγνωση που λαμβάνεται από μια επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνεται επισήμως. Θα πρέπει να ψηφίζει η αρμόδια επιτροπή για να δοθεί εντολή για διαπραγμάτευση σε πρώτη ανάγνωση. Δεύτερον, η εντολή αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και οι συγκεκριμένες υποδείξεις για το τι ακριβώς θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και πού είναι τα όρια αυτής της εντολής. Η εντολή μπορεί να περιλαμβάνει ένα κείμενο ή κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά θα πρέπει να είναι μια σαφής εντολή η οποία θα εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή πριν ξεκινήσει ο εισηγητής τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο. Tiene que haber también un... Τρίτον, θα πρέπει να ψηφιστεί και η σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας. δηλαδή όχι μόνο η εντολή, αλλά και η διαπραγματευτική ομάδα. Ε, ως προς αυτό έχουμε διαφορετικές εμπειρίες, πολύ συχνά πηγαίνουν εσκιώδεις εισηγητές, κάποιες άλλες φορές ε, το προσωπικό των πολιτικών ομάδων, όπως και να έχει όμως η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να υποδείξει ποια είναι η ομάδα διαπραγμάτευσης και ποια είναι η διαπραγματευτική εντολή. Επιπλέον, στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, διαμέσου του Προέδρου της Αρμόδιας Επιτροπής, θα πρέπει οι σκιώδεις εισηγητές και η Επιτροπή στο σύνολό τη θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς προχωρεί η διαπραγματευτική διαδικασία, ποιες είναι οι ενδεχόμενες δυσκολίες και να ζητούνται και συμβουλές ε, ως προς το τι μελιγενέστε με τη διαπραγμάτευση. Και όταν καταλήγουμε σε συμφωνία, η συμφωνία αυτή θα πρέπει να κυρωθεί από την αρμόδια επιτροπή πριν να περάσει στην Ολομέλεια για συζήτηση πιθανών και έγκριση. Ουσιαστικά, τα σημεία αυτά στα οποία μόλις αναφέρθηκα, τα οποία περιλαμβάνονται στον κώδικα δεοντολογίας και περιλαμβάνονται στις συστάσεις ε, του Προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και που περιλαμβάνονται στην επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου στον Πρόεδρο Καζίνη, θα πρέπει να περάσουν στο άρθρο 70 με αναθεώρηση του άρθρου αυτό, ώστε να είναι υποχρεωτικά όλα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή είναι απλώς ε, ε, ηθικό ή πολιτικό καθήκον και τηρούνται ή δεν τηρούνται ε, Στη συνέχεια έχουμε το ρόλο της Ολομέλειας, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει η Ολομέλεια να παρέμβει ώστε να καθορίσει η ίδια την ε, διαπραγματευτική εντολή ή για να τροποποιήσει ή να απορρίψει τη διαπραγματευτική εντολή που έχει ε, καθορίσει η αρμόδια εχει καθορισει η αρμοδια επιτροπη εδώ, όπως γίνεται συνήθως σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν τα δύο άκρα. Αφενός υπάρχουν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να περνούν όλα από την Ολομέλεια, διότι έτσι προσδίδεται ο νομιμότητα σε όλες τις διαπραγματεύσεις, ώστε να είναι το σύνολο των ευρωβουλευτών αυτό που θα έχει δώσει τη διαπραγματευτική εντολή και υπάρχουν αφετέρου αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα βελτιώσει σε καμία περίπτωση την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου, δεν θα επιτρέψει επίσης να κάνουμε διαχωρισμό μεταξύ των υποθέσεων που έχουν μεγάλη σημασία από πολιτική σκοπιά ή μεγάλη σημασία για τη ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και δεν θα γίνεται διαχωρισμό με αυτέ οι οποίε είναι απλώς ε, τεχνικέ αλλαγέ ή δεν ε, προκαλούν καμία διχογνωμία. Θα πρέπει λοιπόν κάπου να γίνει μια διάκριση μεταξύ του ρόλου του Κοινοβουλίου, ε, να δοθεί ένα συγκεκριμένο ρόλος στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, αλλά ταυτόχρονα να την απαλλάξουμε από όλες αυτές τις υποθέσεις που είναι απλώς περιττό άφθος και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ε, στι εργασίε της Ολομέλειας. Στο έγγραφο εργασία που σα παρουσιάζω, παρουσιάζω τρεις τουλάχιστον εναλλακτικέ ε, οδούς που θα μπορούσε ή θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη διαπραγματευτική εντολή, τη σύνθεση της διαπραγματευτικής ομάδας και ούτω καθεξής. Η πρώτη είναι να καθορίσουμε εντολη τη συνθεση της διαπραγματευτικης ομαδας και ουτε θεμάτων που ανάλογα με το πόσο σημαντικά θεωρούνται ή όχι θα πρέπει να περνούν από την Ολομέλεια. Η κατηγορία αυτή των θεμάτων θα πρέπει να είναι περιοριστική, μεν, αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες ε, στο έγγραφο εργασίας. Καταρχάς, οι θέματα, η νομοθεσία που επηρεάζουν ή περιορίζουν απευθείας ε, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών. Δεύτερον, νομοθεσία που τροποποιεί ή που τροποποιεί το συνταγματικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτον νομοθεσία που έχει ε, επιπτώσεις ε, σε πολύ σημαντικό βαθμό για τον προϋπολογισμό, δηλαδή αλλαγές οι οποίες αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό των ε, κονδυλίων για το έτος προϋπολογισμού. Σημαντικές λοιπόν και αδιαμφισβήτητες επιπτώσεις για τον προπολογισμό της Ένωσης. Αυτό που λέει λοιπόν ουσιαστικά το κείμενο είναι ότι όταν το Κοινοβούλιο λαμβάνει ενημέρωση για ένα θέμα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου όταν παραπέμπει στην αρμόδια επιτροπή το θέμα, θα πρέπει ήδη να υποδεικνύει κατά πόσον η έκθεση αυτή, το θέμα αυτό, εμπίπτει σε μία από αυτές τις κατηγορίες και θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετέχει και η Ολομέλεια ε, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Η δεύτερη εναλλακτική οδός θα ήταν να υπάρχουν δύο τουλάχιστον κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες να θεωρούν ότι για το συγκεκριμένο θέμα είναι η Ολομέλεια η αρμόδια για να καθορίσει τη διαπραγματευτική εντολή και τρίτον το 1 δέκατο των ευρωβουλευτών που να ανήκουν τουλάχιστον σε δύο διαφορετικές πολιτικές ομάδες μπορεί να ζητήσουν να αποφασίσει η Ολομέλεια για τη διαπραγματευτική εντολή. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το απλούστερο σύστημα θα ήταν να ανακοινώνεται ότι στην αρχή της επόμενης Ολομέλειας ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα έθετε το ζήτημα της εντολής και να δίνεται ένα περιθώριο 48 ωρών ώστε να λάβουν θέση οι ομάδες ή για να αλλάξει η εντολή, αν υπάρχει εντολή από την Αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια να ψηφίζεται και να ε, αναπέμπεται στην Αρμόδια Επιτροπή ως τροποποιήθηκε ή ως ψηφίστηκε στην Ολομέλεια. Ε, είναι περίπλοκο αυτό το τμήμα, δεν είναι τόσο όριμο ακόμα, είναι πρόημο, ε, ολοκληρώνω, ε, ξέρω ότι μακρηγόρησα, δεν θα ήθελα να καθυστερήσω άλλο για να γίνω σαν το συνάδελφο και φίλο Μιγγελ Άγχελ Μαρτίνεθ. Προτείνω λοιπόν να, γενικώ να μιλώ λιγότερο, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι το θέμα αυτό ουσιαστικά είναι μεταφορά του κώδικα δεοντολογίας στον κανονισμό των περισσότερων από τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχει μια επιτροπή, ένα συζητητής και ούτω καθεξής και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο απλό αλλά και εύκολο ώστε να μπορεί να αποφασίσει η Ολομέλεια χωρίς να παρακολύονται οι εργασίες διαπραγμάτευσης της αρμόδιας επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Ο κύριος Ντάφ τώρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για αυτές τις εξηγήσει. Είναι σημαντικό μου φαίνεται για να απλοποιήσουμε και διευκολύνουμε τις διαδικασίες μας να μην καταλήξουμε να κάνουμε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα και πολύπλοκα από ό,τι ήδη είναι. Αυτό που θέλουμε είναι η διοντολογία που υπάρχει να πραγματοποιείται, να εφαρμόζεται από όλες τις επιτροπές, από όλες τις ομάδες. Γι' αυτό πιστεύω ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί από τη διάσκεψη των πυροέδρων. γιατί πρόκειται για πολιτική απόφαση πρώτης σημασίας. Είναι βέβαια και τεχνικό θέμα αλλά τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι οι πολιτικές διαφωνίες για την πρώτη ανάγνωση πρέπει να εκτιμώνται από τους προέδρους, από τη διάσκεψη των προέδρων. Γιατί θα υποχρεωνόταν έτσι η διάσκεψη να μια στάση πιο στοχευμένη, να δώσει περισσότερη προσοχή δηλαδή, στη γενικότερη κοινοβουλευτική δουλειά του Κοινοβουλίου και ίσως να πρέπει να τους υποχρεώσουμε να διαβουλεύονται και με τους συντονιστές και συντονίστριες. Λίγο παραπάνω, περισσότερο από όσο το κάνουν μέχρι τώρα. εκτιμώ ιδιαίτερα την πρόθεση του κυρίου Γκερέρο να παραμείνει απλός και ρεαλιστής, αλλά σε μια ακόμη ρεαλιστικότερη προσέγγιση θα έπρεπε να αποφύγουμε τον ορισμό κατηγοριών όπως κάνει εκείνος. Αλλά να αφήσουμε το πράγμα στη διακριτική ευχέρεια της διάσκεψης των Προέδρων. Αυτό θα ήταν νομίζω το καλύτερο. Τέλος, ερωτώ. Γιατί στην Ολομέλεια προτείνεται να ισχύει πάντοτε η απόλυτη πλειοψηφία. Συνήθως η απλή πλειοψηφία αρκούσε. Και να ζητάμε απόλυτη πλειοψηφία στις αρχές μιας διαπραγμάτευσης μου φαίνεται κάτι πολύ δύσκολο. Δεν μπορούμε πάντοτε από την αρχή μιας νομοθετικής διαδικασίας να πετύχουμε τόσο μεγάλη διακομματική συνεργασία. Πολλές, σε πολλές περιπτώσεις μια απόφαση της Ολομελίας μπορεί να είναι μεταξύ της σχετικής και της απόλυτης πλειοψηφίας, της απλής και της απόλυτης πλειοψηφίας. κάτι τέτοιο θα αποδυνάμωνε αν το απαγορεύαμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μακντάφ Πολύ δύσκολο θέμα. Πρέπει να υπάρξει μια δύσκολη βέβαια εξισορρόπηση. γιατί θέλουμε η διαδικασία να είναι απλή και κατανοητή, αλλά απ' την άλλη θέλουμε και μεγαλύτερη δημοκρατική, μεγαλύτερο θεμητό χαρακτήρα εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί η διαδικασία που ακολουθούσαμε μέχρι τώρα επιτάχυνε μεν τα πράγματα αλλά μείωνε την δημοκρατική νομιμότητα. Οι περισσότεροι δεν μπορούν καν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες. Στη συνθήκη της Λισαβόνας ένας από τους στόχους είναι η απλοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Φοβόμαστε λοιπόν μήπως δημιουργηθεί ένα σύστημα ακόμη πιο πολύπλοκο από ό,τι μέχρι τώρα και δυσνόητο. Η ιδέα να μπορούμε να περάσουμε την πρώτη ανάγνωση πολύ γρήγορα ήταν να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά ο κίνδυνος είναι μήπως οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπως λένε ορισμένες συστάσεις αποδυνάμωσης μπροστά στο Συμβούλιο, ενώπιον του Συμβουλίου έναντι του Συμβουλίου. Εσείς βέβαια έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από μένα, αλλά και διαβάζοντας απλώς πώς ήταν τα πράγματα το 90, βλέπω ότι το Κοινοβούλιο σε μερικές περιπτώσεις ήταν διηρημένο και γι' αυτό εποφελούνταν το Συμβούλιο και μας αγνοούσε ή γενικά είχαμε αποδυναμωμένη θέση. Πρέπει λοιπόν όσο το δυνατόν περισσότερο να δημιουργούμε ενωμένα μέτωπα. Φοβάμαι ότι αν εγκρίνουμε αυτού του είδους την προκαταρκτική αποδοχή των εντολών γρήγορα, ότι θα αποδυναμωθούμε και σε ορισμένα θέματα θα υπερισχύσει το πολιτικό ένσυτικτο. γιατί μερικές προτάσεις είναι πολύ δυσνόητες και πρέπει να τονίσουμε την πραγματικότητα και όχι τις πολιτικάντικες διαδικασίες. Ξέρω ότι όλα αυτά γίνονται για μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα και διαφάνεια, αλλά έχω αμφιβολίες. Θέλω λοιπόν να πω ότι πολλοί ε, αισθάνονται κάποια απογοήτευση γιατί γιατί ούτε η Ολομέλεια ούτε καν η Επιτροπή δεν καταλαβαίνουν καμιά φορά που πάνε τα πράγματα στη διαπραγμάτευση. Το θέμα λοιπόν δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν πληροφορείται η Ολομέλεια, αλλά ούτε καν η Επιτροπή μας. πάνε στον τριμερή διάλογο οι εισηγητές και οι εισηγήτριε και δεν γίνεται καμία διαβούλευση με την Επιτροπή μας. Έχουμε μπροστά μα τελεσμένα γεγονότα. Ενώ ο δικός μας ρόλος, όχι ολομέλεια, είναι γενικά η έγκριση όλων αυτών. Λέω λοιπόν ότι το θέμα είναι αμφιλεγόμενο. Πώς θα καταλήγαμε δηλαδή στην ιδεώδη εξισορρόπηση. Δεν έχω καμία πρόταση να κάνω, αλλά πρέπει να το ξαναδούμε. Αν πρέπει να καθορίσουμε τέτοιες κατηγορίες ή να αφήσουμε τα πράγματα στη διακριτική ευκαιρία της διάσκεψης των Προέδρων. αλλά σε όλους εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αρμόδια επιτροπή κάθε φορά είναι το σημαντικό θέμα όμως και πρέπει να, δεν πρέπει να αποδυναμώνουμε τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Ακόμη και αν αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη διαφάνεια. Σας κατευχαριστούμε. Μέντες Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω να συγχαρώ καταρχάς τον κύριο Γκερέρο για την παρουσίαση που μας έκανε. όχι τόσο μεγάλη όσο αυτή που μας κάνει συνήθως ο κύριος Μαρτίνεθ, αλλά εις βάθος όπως μα μας κάνει και ο Αντιπρόεδρος και νομίζω ότι ε, έθεσε το θέμα στα σωστά του πλαίσια και μάλιστα και το έκανε και με το σωστό πνεύμα ε, συνεργασία, ζητώντα από όλου συνεργασία και ξεκινώντα τη συζήτηση για μία απόφαση η οποία θα πρέπει να είναι με τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Συγχαρητήρια λοιπόν, ε, διότι ε, παρουσίασε ένα έγγραφο εργασίας με μεγάλη οριμότητα. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε ενώπιον μια εξ αυτών των περιπτώσεων που οι εμπειρογνώμενες ονομάζουν ε, μετατροπή των πραγμάτων. Ε, παλιά είχαμε τρεις αναγνώσεις ή συνδιαλλαγή. Και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία μας παρουσίασε ο κύριος Γκερέρο για τον αριθμό των συμφωνιών ε, στις οποίες καταλήξαμε σε πρώτη ανάγνωση, το 70% λέει πολλά. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, ένας διαρθρωτικός λόγος. Το Κοινοβούλιο, όπως είπε και ο κύριος ε, Τρασκόσκι, ε, είχε δυσκολίε για να έχει κοινέ θέσει στη δεκαετία του 90. Υπάρχει όμως και, ένα ακόμα, και ένας ακόμα λόγος και γι' αυτό πριν είπα ότι είναι διαρθρωτικός. Για να παρουσιάσει κάποιο τροπολογία σε δεύτερη ανάγνωση απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο κατανόησε ότι το καλύτερο είναι να υπάρχει ε, η ευρύτερη δυνατή συνένεση σε μια ε, θέση εξ αρχής. Αν δείτε τα θέματα τα οποία έφτασαν σε δεύτερη ανάγνωση και που πέρασαν και τροπολογίες σε δεύτερη ανάγνωση, θα δείτε ότι είναι ελάχιστες τροπολογίες. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι αν πρέπει να νομοθετήσουμε και δώσαμε και μάχη για να νομοθετούμε περισσότερο, οποιαδήποτε αλλαγή για τη συνθήκη σημαίνει περισσότερες αρμοδιότητες και περισσότερη εξουσία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξουσία. Και προέκυψε κάτι το οποίο δεν ήταν μεν γραμμένο σε συνθήκες, αλλά ε, είναι η διαρθρωτική λογική, διότι είναι πολύ πιο απλό να καταλήξουμε σε συμφωνία εκ των προτέρων παρά εκ των υστέρων. Και επιπλέον, οι νομοθετικές ε, λύσεις που απαιτούνται από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, θα πρέπει να γίνονται ταχύτατα. Δεν μπορεί να συζητάμε για μήνες και για χρόνια θέματα τα οποία απαιτούν γρήγορη απάντηση. Όλο αυτό ο κόσμο των νέων τεχνολογιών, όπου όλα είναι ταχύτατα και άμεσα θα πρέπει ε, να συνοδεύονται και από νομοθετικό έργο το οποίο είναι προσαρμοσμένο σε αυτή τη ταχύτητα. Mm. Επομένως υπάρχει πολιτική ανάγκη και, επομέν, και σε αυτήν ανταποκρινόμαστε. Αν εγκρίνουμε σε πρώτη ανάγνωση λοιπόν, ανήκουμε στον πραγματικό κόσμο και νομοθετούμε βάσει της πραγματικότητας. Πρόκειται λοιπόν για μια λογική μετατροπή, αξία αξιέπαινη μετατροπή. Mm-hmm. Ε, στην πολιτική μου ομάδα συζητήσαμε το θέμα και κάποιοι έλεγαν όχι, όχι, πρέπει να απαγορεύονται οι συμφωνίες σε mm. πρώτη ανάγνωση. Μα θα τις απαγορεύσουμε η ανάγνωση γίνεται για να επιτύχουμε συμφωνία. Αν συμφω... επιτυχάνουμε συμφωνία νωρίτερα, γιατί να κάθεσαι να συζητάς ε, ε, περαιτέρω διαδικαστικά στάδια χωρίς λόγο. Θεωρώ ότι είναι λογικό και είναι και καλό, θετικό και βρίσκεται και στη φύση των πραγμάτων, αν μου επιτρέπετε. Το λέω εγώ ως νατουραλιστής. Θα πρέπει λοιπόν λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, να κάνουμε και μία απόπειρα να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και πιο διάφανη. Διότι υπάρχει δυνατότητα ε, να παρουσιαστούν όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας ανέφερε και ο κύριος Γκερέρο. Να ε, μην μαθαίνουν οι συναδελφοί τι συμβαίνει, να είναι λίγο ε, και καλυμμένα τα πράγματα και να βρίσκονται ε, πρωτετελεσμένου οι συνάδελφοι. Ο καθένας όμως βλέπει τη συμφωνία από την πείρα του. Εγώ μόλις ε, τελείωσα τη συμμετοχή μου σε μία μακροσκελέστατη διαπραγμάτευση, η οποία τελικώς κατέληξε σε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και πρέπει να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο οι πρόεδρος της Επιτροπής, οι συγητές, οι σκιώδεις συγητές αντιμετώπισαν το θέμα είναι παραδειγματικός τα τέσσερα βασικά ζητήματα τα οποία συζητώνται στον κώδικα δεοντολογίας τηρήθηκαν κατά γράμμα. Και συνεχώς ενημερωνόμασταν όλοι οι συγητές και οι συγητές, μας δίνανε πληροφορίες, η Επιτροπή, οποιοδήποτε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λοιπόν ο οποίος μπορεί να βρει ψεγάδι στον τρόπο με τον οποίο τηρήθηκε η διαδικασία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι να μεταφέρουμε αυτό τον κώδικα διοντολογίας στον κανονισμό ώστε να είναι υποχρεωτικό. Επιμένω ότι από την πείρα μου τα σημεία τα οποία ανέφερε ο κύριος Γκερέρο ε, φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διεξάγονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι το ουσιώδες. Και μου δόθηκε εντύπωση στις παρεμβάσεις που άκουσα μετά από τα όσα είπε ο κύριος Γκερέρο ότι χάνουμε το στόχο μας ουσιαστικά. Βλέπουμε τις λεπτομέρειες και χάνουμε το στόχο μας. Να σας πω γιατί. Ε, κατά την άποψή μου, ε, δεν επικεντρώσαμε επαρκώς τη συζήτηση στο τι γίνεται αν κάποιος δεν τηρεί την εντολή του, ας πούμε. Να τα βάλουμε στη σωστή ε, διάσταση. Το πιο σημαντικό είναι αυτοί οι κανόνες του κώδικα διοντολογίας να μεταφραστούν σε κανονισμό. Το άλλο είναι ίσονο σημασία. Νομίζω, όπως και ο εισηγητής, ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να οριμάσουν και γι' αυτό πρέπει να γίνει συζήτηση. Και θεωρώ λοιπόν ότι το να καθορίσουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα ή κάποιες νομοθετικές προτάσεις λόγω περιεχομένου, οι οποίες θα πηγαίνουν οπωσδήποτε στην Ολομέλεια, μου φαίνεται ότι δημιουργεί κάποια προβλήματα. Πρώτον, ο σαφής ορισμός των θεμάτων αυτών και δεύτερον, ότι μπορεί να είναι πολύ σημαντικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι θέματα στα οποία δεν υπάρχει διάσταση απόψεων. Επίσης υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα στοιχεία που μας ανέφερε ο κ. Γκερέρο, όπως για παράδειγμα το REACH. Το REACH δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχουμε για να πάνε οπωσδήποτε στην Ολομέλεια. Αλλά είχαμε μια παθιασμένη συζήτηση με πάρα πολλέ επιπτώσει κάθε μορφή ε, για το REACH. Εάν λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος προτάσεων ε, για τις οποίες η διαπραγματευτική εντολή ε, θα πρέπει να λαμβάνεται στην Ολομέλεια, ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οριμάσει. Αυτός πρώτο στοιχείο. Δεύτερον, για την Ολομέλεια. Άκουσα πολλούς συναδέλφους να λένε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να ενημερώνονται σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαπραγμάτευση, ποια είναι η εντολή και το καθεξής. Αμφιβάλλω αν θα είναι αποτελεσματικό αυτό. Εγώ ως μέλος ε, του Κοινοβουλίου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σας το λέω σαφώς. Απ' τη μια δημοσιοποιείται το θέμα περισσότερο, αλλά δεν είναι απαραίτητο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτό. Διότι η αποτελεσματικότητα και εκεί που συναντιούνται αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα το ζήτημα είναι τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής. Αυτοί είναι αυτοί που γνωρίζουν τι συζητιέται και αυτοί μπορούν να κάνουν και τη διάκριση ε, με επιχειρήματα για το περιεχόμενο της εντολής. Στην Ολομέλεια, εγώ να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι δεν είναι πιο αποτελεσματικά τα πράγματα θα είναι μια τυπική διαδικασία ε, και από τη μια θα είμαστε ικανοποιημένοι από πλευράς προβολής ενός θέματος, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι ε, θα έχει ε, απτές συνέπειες όταν ε, θέλουμε να αναγνωρίσουμε τα θέματα αυτά. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να το ξανασκεφτούμε αυτό το ζήτημα. Εξακολουθώ να θεωρώ ότι η αρμόδια επιτροπή είναι αυτή η οποία γνωρίζει καλύτερα ένα ζήτημα και εκεί μπορούν να συζητηθούν και τα πολιτικά ζητήματα, τα οποία είναι και αυτά τα οποία θα ισχύσουν όταν θα δούμε αν θα εγκρίνουμε ή θα κυρώσουμε ή θα απορρίψουμε μια εντολή. Γνωρίζω τι ικανότητες έχουν οι πρόεδροι των επιτροπών και πόσο επαγγελματίες είναι. Το περιθώριο ευελιξία σε τεχνικό επίπεδο, αν μου επιτρέπετε, είναι σπάνιο. Υπάρχουν και πολιτικά συμφέροντα απόλυτα ένομα. Επομένως, εκεί που μπορούν να αποφασίσουν καλύτερα, κατ' εμέ, είναι στην αρμόδια επιτροπή. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να λαμβάνεται απόφαση. Κύριε Πρόεδρε, Αυτές όμως είναι σκέψεις οι οποίες προέκυψαν εν θερμό ακούγοντας ε, τα όσα συζητούνται εδώ. Γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους, να ακούσω τι έχουν να συνεισφέρουν και να αφήσουμε, όπως είπε και ο εισηγητής, να οριμάσει λίγο το θέμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ε, να συνειδητοποιήσουν και οι πολίτες την αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως το αντιπροσωπευτικό όργανο που ενδιαφέρεται για τα θέματα που τους αποσχολούν και που θέλει να τους τα επιλύσει το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε τον κύριο Μεντετεβίγο. Νομίζω ότι έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Χέφνερ τόδο. Εγώ πρέπει να λείψω ένα τεταρτάκι. Θα ζητήσω από τον κύριο Ταρκόσκι να αναλάβει τα ημεία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνω μία απόπειρα να μην πω στον όλο ανταγωνισμό για το ποιος θα μιλήσει πιο πολύ. Μάλιστα θα ήθελα να εξαιρεθώ από αυτό το ανταγωνισμό. Φυσικά κατανοώ το γεγονός ότι εδώ με το έγγραφο αυτό ξεκινάμε και δεν κλείνουμε μια συζήτηση. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να μιλήσουν όλοι για όλες τις πτυχές του κειμένου η δική μας, η δική μου κατεύθυνση στο θέμα αυτό είναι η εξής. Η δημοκρατία ζει από την ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά σκοπός πάντα είναι να λαμβάνονται αποφάσεις όσο δυνατόν γίνεται με ελευθερία λήψεως αποφάσεων όχι με περιορισμό αυτή τη λήψη αποφάσεων. Άρα, πώ θα οργανώσουμε, θα διοργανώσουμε τον τρόπο λήψη αποφάσεων. Το κοινοβούλιο αυτό έχει και χρειάζεται, θεωρώ, ένα ολόκληρο πλωστάσιο για, σε ό,τι αφορά την λήψη αποφάσεων, σε ό,τι αφορά την συναπόφαση με άλλα θεσμικά σώματα και θεωρώ ότι είναι θετικό σε ό,τι αφορά την εκλογή, την επιλογή του εκάστοτε κατάλληλου μέσου, να μην περιοριστούμε. Υπάρχουν πολλά μέσα. Καταρχάς, ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να συντείνουν υπέρ μιας ε, απόφαση σε πρώτη ανάγνωση, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να μην αποτελεί τον πλέον κατάλληλο τρόπο για την λήψη της εκάστοτε απόφασης. είτε πρόκειται για τον προπολογισμό, είτε πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά τα κριτήρια δεν μπορούμε να τα ορίσουμε με ακριβείς τρόπους όταν για παράδειγμα επηρεάζονται θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Κατά πόσον αυτό περιλαμβάνει όλες τις εκτέσεις της Επιτροπής ΛΥΠΕ και ποιος αποφασίζει αυτός. Εγώ, κοιτάξτε, αυτό που με ανησυχεί είναι να μπούμε στην διαδικασία να βρούμε τελικά μια φαινομενική λύση για θέματα τα οποία τελικά χρήζουν πολιτικής απόφασης και νομίζω ότι αυτή η πολιτική απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται εκεί που υπάρχει η καλύτερη αρμοδιότητα ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε ζητήματος. Γι' αυτό λοιπόν είμαι ιδιαίτερα σκεπτικός και επικριτικός σε ό,τι αφορά την κατηγοροποίηση της σύσταση ενός καταλόγου και επίσης σε ό,τι αφορά την ε, διαδικασία. Θα ήθελα να αναφέρω ότι είμαι και, και μάλλον επικριτικός για το θέμα του γιατί να χρησιμοποιηθεί απόλυτη πλειοψηφία ενώ πολύ πιο σημαντικά θέματα τα αποφασίζουμε με απλή πλειοψηφία. Δεν έχω πιστεί, αλλά κοιτάξτε, τώρα ξεκινάει η διαπραγμάτευση και, εν πάση περιπτώσει, εγώ δηλώνω ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν διαπραγματεύσει. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, κανείς άλλος μετά το λόγο. Ο κύριος Κέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ από τα όσα άκουσα θα ήθελα καταρχάς να κάνω μια προκαταρκτική δήλωση. Έλεγα πριν ότι πριν να ετοιμάσω ένα σχέδιο έκθεσης ήθελα να κάνω ένα έγγραφο εργασία ακριβώς για να δω λίγο πού βρίσκονται οι διαθέσεις σας, οι προτάσεις σας και οι θέσεις και ημών των συντονιστών και των σχεδόν εισηγητών και των μελών της Επιτροπής μας. Αυτό που αντλώ δίδαγμα από τη σημερινή συνεδρίαση, δεν ξέρω αν όλοι όσοι είμαστε εδώ αντιπροσωπεύουμε όλο το φάσμα των μελών, αλλά αντιλαμβάνομαι κάτι το οποίο ήδη γνώριζα. Ναι. Και αυτό είναι ότι το ουσιώδες είναι στο άρθρο 70 να περάσουν αυτά που έχουμε στον κώδικα διοντολογία. Αυτό είναι η ουσία. Το δεύτερο ουσιαστικό σημείο είναι ότι το αποφασιστικό κομμάτι πέρα από ε, με την εξαίρεση συγγνώμη, συγκεκριμένων περιπτώσεων είναι να λαμβάνονται αποφάσεις από την αρμόδια επιτροπή διότι αυτές γνωρίζουν τα διάφορα ζητήματα και τρίτον όπως είπε και ο κύριος Τρασκόσκι οι εντολές δεν μπορεί να είναι συγκεκριμένες κλειστές εντολές οι οποίες δένουν τα χέρια των διαπραγματευτών ε, στη διαπραγματευσή τους με το Συμβούλιο. Ε, αυτό επαφείται σε κάθε επιτροπή. Υπάρχουν επιτροπές οι οποίες όταν καθορίζουν τη διαπραγματευτική εντολή μπορεί να ετοιμάζουν μια γενική εντολή με κάποιες γενικές κατευθύνσεις και κάποιες άλλες επιτροπές μπορεί να καθορίσουν μια εντολή πολύ πιο συγκεκριμένη, αλλά θα πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί. Αν είναι πολύ συγκεκριμένη μια εντολή, δεν θα πρέπει να αποδυναμώνει την ε, διαπραγματευτική μας θέση. Δηλαδή, ε, να, ή να να μην επιτρέπει να είμαστε πιο ευέλικτοι. Αυτά λοιπόν εν είδη πρώτων συμπερασμάτων. Το άρθρο 70 θα πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του κώδικα διοντολογίας. Στο επίκεντρο θα πρέπει να βρίσκεται η αρμόδια επιτροπή και θα πρέπει να υπάρχει και κάποια ευελιξία για τη διαπραγματευτική εντολή. Δεύτερο τώρα, το οποίο λαμβάνω ως αρνητικό μάθημα, οι κατηγορίες ε, θεμάτων δεν φαίνεται να δημιουργούν και μεγάλο ενθουσιασμό, τουλάχιστον από τις παρατηρήσεις που άκουσα από τα μέλη της Επιτροπής. Θα πρέπει να το ξαναδώ, αλλά να το ξαναδώ γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι ε, είναι περιορισμένος ο ενθουσιασμός επί του θέματος. Τρίτον, το να χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία αν περάσει ένα θέμα στην Ολομέλεια δημιουργεί προβλήματα. Εγώ συναντήθηκα με τον κύριο Λένε. Ο κύριος Λένε ήδη μου το έθεσε το θέμα αυτό, αλλά όταν μου το έθεσε ήδη ήταν έτοιμο το έγγραφο εργασίας. Είχα όμως λάβει υπόψη και το ενδεχόμενο να μην είναι και τόσο καλή λύση αυτή η απέτηση να υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Υπάρχει λοιπόν πεδίο συμφωνίας εάν επιλύσουμε το θέμα της Ολομέλειας. Πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τι ρόλο διαδραματίζει η Ολομέλεια, πότε τον διαδραματίζει, εάν πρέπει να τον διαδραματίσει σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, εάν πρέπει να αποφασίζει μόνο όταν ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής ε, θέσει το ζήτημα στη διάσκεψη των Προέδρων και η διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσει να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια, που είναι ε, η πλέον απλουστευμένη διαδικασία, ε, με βάση και τα όσα έλεγε ο κύριος Νταφ. Με βάση αυτά λοιπόν, όπως σας είπα, με την ησυχία μου θα ετοιμάσω ένα σχέδιο έκθεσης, το οποίο θα είναι πλέον μια συγκεκριμένη πρόταση. Είμαι πάρα μα πάρα πολύ απογοητευμένος διότι απουσιάζει ο κύριος Μέντες Δεβίγο. Για αυτούς που δεν είναι Ισπανοί, αναφέρθηκε στον κύριο Ραχόη, που είναι ο υποψήφιος του Λαϊκού Κόμματος στις εκλογές στην Ισπανία, ε, τον οποίο ανέφερε ως συνταγματολόγο και με κάποιο και καλυμμένο τρόπο αναφέρθηκε και στο Μοντεσκέ, διότι είπε ότι οι νόμοι είναι οι απαραίτητες σχέσεις που προκύπτουν από τη φύση των πραγμάτων. Το να συγκρίνουμε λοιπόν το Ραχώη με το Μοντεσκέ νομίζω ότι είναι ε, υπερβολή και λίγα λέω. Στην ουσία όμως η παρέμβασή του ήταν όλα όσα εξέλεβα, να επικεντρωθούμε δηλαδή ουσιαστικά στην ε, μεταφορά του κώδικα διοντολογίας στο άρθρο 70 και να σκεφτούμε λίγο καλύτερα ή πολύ καλύτερα το πώς ε, θα λαμβάνει θέση η Ολομέλεια εάν απαιτείται και ποια είναι η πιο απλή διαδικασία για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Allora, ε, ωραία, δεν έχουμε άλλε παρεμβάσει. Ζητώ συγγνώμη για τη σύντομη απουσία μου. Ε, και νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε τι προθεσμίε για να μπορέσει να ετοιμάσει και ο εισηγητή το σχέδιο έκθεσή του. 21 Νοεμβρίου είναι καλή ημερομηνία, ώστε να μπορέσουμε να ψηφίσουμε στις 26 Ιανουαρίου στην Επιτροπή. Ωραία. Η έκθεση Γκουρμάη έχει αναβληθεί για αύριο. Επομένως, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και η συνεδρία συνεχίζεται αύριο στις 9.30, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρο, στι 9 ακριβώ αύριο. Αλλά πρέπει να γίνει συνεδρία των συντονιστών τώρα. Παρακαλώ λοιπόν οι συντονιστέ να παραμείνουν στην αίθουσα.